Στην, ε, στο ροστάσιο της, BM, της BMW και να τους πει ότι εγώ θέλω τόσο πολύ αυτή τη συμφωνία που δεν με νοιάζει για τις δουλειές σας. Το έκανε αυτό ο κ. Φαράτζ. Αυτό θα ήταν το έντιμο να πράξει. Ο Δόκτωρ Λίαμ Φόξ άραγε είπε ποτέ ή έλεγα παλιότερο θα είναι η πιο εύκολη εμπορική συμφωνία στην ιστορία μας, αλλά τελικά βλέπω ότι είναι πιο περίπλοκο από ό,τι είχα υποσχεθεί πριν το δημοψήφισμα. Ο Μπόρις Τζόνσον, άραγε, πήγε στους γιατρούς και τι νοσοκόμε του Εθνικού Συστήματος Υγεία να τους πει ότι ναι, σας είχε υποσχεθεί 350 εκατομμύρια ε, λίρες τη βδομάδα έξτρα προπολογισμό, αλλά τελικά λυπάμαι πάρα πολύ, δεν τα καταφέρνω. Το έκαναν αυτό. Ειλικρινά. Για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, θα έπρεπε να δείξουν λίγη μετριοφροσύνη για λίγη μετριοπάθεια. Λίγη ταπεινότητα. Επίσης πιστεύω, ναι, ε, ε, μου πέδειξαν μια έκθεση της κυβέρνησης που δημοσιεύτηκε πέρσι τον Νοέμβρη, της Βρετανικής κυβέρνησης, που έλεγε ότι ε, το κόστος ε, μιας ε, Αποχώρηση χωρί συμφωνία θα ήταν 9,3% του ΑΕΠ. Είσαστε έτοιμοι, είσαστε πρόθυμοι να πληρώσετε αυτό το, τίμημα. Είσαστε πρόθυμοι να θυσιάσετε όλες αυτές τις ε, θέσει εργασία για αυτό το όνειρο της κυριαρχίας, τη δίθεν κυριαρχίας. Τι θα φέρει για εσά αυτό το όνειρο. Κύριε Κόμπερν, παρακαλώ πολύ, λέει η πρόεδρος. Συγγνώμη, μισό λεπτό κύριε Αντιπρόεδρε, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Κύριε Κόμπερν, εμείς οι δύο έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Ε, εγώ είμαι ιδιαίτερο, ιδιαίτερο, δεν ξέρω εσείς τι είστε. Παρακαλώ πολύ, μη διακόπτετε. Παρακαλώ πολύ, ακούστε, ακόμα και αν διαφωνείτε, ακούστε με σεβασμό και ίσως να μάθετε κάτι. Κύριε Πρόεδρε, εγώ άκουσα, τον κύριο Κόλμπερν και λέει η ελευθερία είναι πιο σημαντική. Ε, οπότε, γιατί δεν έχετε το θάρρο, δεν δείχνετε το θάρρο να πάτε στο Σάντελαρτ, να μιλήσετε με του εργάτε τη Νισάν. Πηγαίνετε στο, στην Οξφόρδη να μιλήσετε με τους εργάτες του εργάτε του, εργοστασίου που βγάζει τα μίνι, τη BMW κλπ. Πηγαίνετε και στην Ιρλανδία. Πηγαίνετε εκεί όπου από το 98 ε, εξαφανίστηκε η βία και βασιλεύει η ειρήνη. Γιατί δεν λέτε ότι το δικό μου όνειρο είναι πιο σημαντικό από τη δική σας ειρήνη και θα δεχτώ ένα σκληρό σύνορο αν αυτό μου επιβεβαιώνει τις προσδοκίες μου για ένα ε, Brexit χωρίς συμφωνία. Γνωρίζετε τι σημαίνει 16,9 εκατομμύρια εγώ πάντα ακούω το 17,4 εκατομμύρια, αλλά το 16,1 εκατομμύρια είναι επίσης Βρετανοί πολίτες που ψήφισαν να παραμείνουν. Δεν εξαφανίστηκαν. Και η ουσία της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας δεν είναι να σεβόμαστε για τη θέση των δημοψηφιών στις χώρες μας. Δεν είναι ουσία, πεμπτουσία της Δημοκρατίας να προσπαθούμε να χτίσουμε γέφυρες και να βρούμε λύσεις δεν θα έπρεπε αυτό να είναι το επόμενο βήμα μας. Και να είμαι πολύ σαφής. Γιατί η Κομισιόν επιμένει τόσο πολύ για την ακαιρεότητα της εσωτερικής αγοράς. Γιατί δεν λέμε ας ανοίξουμε τα σύνορα. Να σας πω το εξής, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν για κάποιο λόγο το Ενωμένο Βασίλειο αποφάσιζε να συνάψει εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, με τους δικούς τους όρους, Τα κοτόπουλα με χλωρίνη θα μπαίνουν στο Ενωμένο Βασίλειο. Ε, εμείς δεν θέλουμε να πούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο όμως ε, πώς θα προστατεύσει τον εαυτό του. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη δική μας αγορά. Γι' αυτό το λόγο ε, δεν έχουμε φυστεί προσπαθειών. Ε, επουδενή να προσπαθήσουμε να ε, συμφιλιώσουμε τις κόκκινες γραμμές της κυρίας Μέη με την με το δικό μας ε, καθήκον να προστατέψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ακαιρότητα τη ε, εσωτερική αγοράς. Η συμφωνία αποχώρηση που υποβλήθηκε, που παρουσιάστηκε, είναι η μόνη λύση που μπορεί να εξασφαλίσει αυτό. Αυτή είναι μια θέση που στηρίζει η Κομισιόν εκ μέρους όλων σας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για να προστατεύουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών είτε ζουν στην υπηρετική Ευρώπη είτε στον Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμανς. Η κυρία Τσιώτα από το Συμβούλιο έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις που κάνετε, για τα σχόλιά σας. Θα ενημερώσω δεόντω τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι σαφέ ότι πιέζει πάρα πολύ το ζήτημα του Brexit, ιδίω για τη σύνοδο τη επόμενη εβδομάδα. Ήδη αντιμετωπίζουμε τι άμεσε συνέπειε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τι στρατηγικέ προκλήσει που θα καθορίσουν το κοινό μα μέλλον τα επόμενα χρόνια. Στο πνεύμα λοιπόν αυτό, τα διαφορετικά ζητήματα τα οποία προβλέπονται και τα οποία συζητήσατε ουσιαστικά θα αποτελούσουν μέρος της επόμενης ευρωπαϊκής στρατηγικής ατζέντα. Θα έχουμε το επόμενη, την επόμενη άτυπη σύνοδο που θα μας δώσει την δυνατότητα να θέσουμε το μακροπρόθεσμο αυτό θεματολόγιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κυρία Τσιότ. Ολοκληρώνει στο σημείο αυτό η συζήτηση. Buongiorno. Καλημέρα σας. Ας ξεκινήσουμε τις ε, ψηφοφορίες. Καθίστε παρακαλώ πολύ, ετοιμαστείτε. Παρακαλώ. Dear colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από ένα χρόνο εγκρίναμε μια τοποθέτηση όσον αφορά τον κανονισμό ειδών διτής χρήση που περιορίζει τον, την εξαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων σε δικτατορικά καθεστώτα και διευκολύνει επίσης τα προϊόντα κρυπτογράφησης και ταχθήκαμε 92% υπέρ τη πρόταση αυτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτο δικαίου, που πλήττονται παντού στον κόσμο. Νέε δικτατορίε τώρα στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή αναπτύσσονται, αναδύονται και παλαιότερε όπω ε, η Κίνα γίνονται όλο και πιο κατασταλτικέ στην στάση του. Έχουμε πραγματικά τραγικέ καταστάσει όπω με τον δημοσιογράφο Κασόγκη, ο οποίο ε, δολοφονήθηκε, κάθηκε, ε, ε, διαμελίστηκε από το καθεστώς οδική Αραβίας. Χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο τέτοιες τακτικές και τα εγκλήματα αυτά γίνονται όλο και πιο α, διαδίδονται όλο και περισσότερο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς να συνειδητοποιήσουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την διαδικασία αυτή για λόγους ασφάλειας αλλά και λόγους ηθικούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τους πολίτες παντού στον κόσμο που θέλουν να βελτιώσουν την κοινωνία, που λένε την αλήθεια απέναντι στην εξουσία, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ζουν σε καθεστώς ελευθερίας και ασφάλειας. Εμείς προσπαθούμε να προασπίσουμε τις βασικές μας αρχές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όμως φαίνεται διαφορετικό και αρνήθηκε να εγκρίνει μια κοινή θέση προκειμένου να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για το θέμα αυτό. Ιδίω έγινε μια τελευταία αλλαγή στη στάση του κυρίου Μακρόν, του ίδιου του κυρίου Μακρόν, που σταμάτησε τελικά διαδικασία. Η Γαλλία, η Σουηδία, η Φιλανδία και άλλα κράτη-μέλη θεωρούν τελικά ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει και αυτές να συμμετέχουν ανυπέτειες για τα εγκλήματα αυτά, κερδίζοντας παράλληλα. Καλό λοιπόν το Συμβούλιο να ακούσει προσεκτικά όλες τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πραγματικά να θέσει τις αξίες μπροστά από το κέρδος. Λοιπόν, ας ψηφίσουμε τώρα την έκθεση αυτή, καθώς επίσης και όλες τις υπόλοιπες διασφαλίσεις εγγύησης κατά του σκληρού Brexit. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπούκνερ. Σας έδωσα το λόγο να αφορά την έκθεσή σας, την οποία τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Μιχαήλοβα. Μονομαστική κλίση. Άρχιτη ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Ζροντεύσκη. Μονομαστική κλίση, άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Σλοτόφσκι τώρα. Με ονομαστική κλίση, άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Φωτίγκα. Με ονομαστική κλίση. Άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Έκθεση Φωτίγκα όσον αφορά την Συμφωνία Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφγανιστάν. Τροπολογία παριθμών 1. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 48 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση άρθρη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπερθμών 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μονομαστική κλίση το ψήφισμα στο σύνολό του άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Μακοβέη, μονομαστική κλίση, άρτη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση Βάουτμανς. Όσον αφορά τους ειδικούς αντιταλμένους Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει καμία γραπτή αντίρρηση αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη συντήρηση αυτή. Για να ακολουθήσουμε όμως το άρθρο 13, παράγραφος 16, θεωρείται ότι έχει εγκριθεί η σύσταση αυτή. Τώρα, έκθεση Λόκεγκάρτ, μονομαστική κλίση, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο η πρώτη αναγνώση του Κοινοβουλίου. Έκθεση Κοέλιο τώρα. Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής, όλες μαζί υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 252 τροπολογία εγκρίνονται οι προηγούμενες. Ηλεκτρονική επαλήθευση, σας παρακαλώ πολύ. Ηλεκτρονική επαλήθευση για να δούμε το πραγματικό αποτέλεσμα. Άρτη ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνονται. Ναι, ναι, κάνα λάθος, συγγνώμη. 252D, με κλίση, άρτη ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρασε. Απορρίπτεται. 253 πρώτο τμήμα μονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα μονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 254D με ονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 235-241 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Το σύνολο τώρα κειμένου με ονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται κατά αυτόν τον τρόπο εκλοκληρώνεται την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έκθεση Ντάλι, τροπολογίε τη καθήλυνα αρμόδια επιτροπή ψηφίζουμε από κοινού υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνονται. Τροπολογία 1, μονομαστική κλίση, άρτη ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 σε 4 τμήμα πρώτα Πρώτο τμήμα άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Με ονομαστική κλίση. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 19. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ήταν πολύ δύσκολο ουσιαστικά να δούμε το αποτέλεσμα. 24 τώρα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση όσον αφορά το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 24. Πολύ ωραία, έρθει ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Και εδώ με μικρή διαφορά. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Πρώτο τμήμα. Άρθρη ψοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 32. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 37. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 49, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 49, άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρθιψη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 57. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η Ηλεκτρονική επαλήθευση, άρτη, άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση και για το τμήμα αυτό, άρτη ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 60, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 68 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 73 πρώτο τμήμα, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 80. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 82 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση άρθρη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 92 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 104 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της 104 άρτη ψηφοφορία.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 εγκρίνεται. 140 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. 168 υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. 169 υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. 176 υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. 177 υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 184 σε ε, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 186. Άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 216 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 224 υπέρ κατά Αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος, άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 232 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 261 δι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Καταπίπτει η 262, 70-71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Καταπίπτει 263, 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 264. Πάμε στην 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 76 άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 252, τροπολογία 77, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 253, τροπολογία 93, πρώτο τμήμα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κατά πίπτη 254, τροπολογία 103, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. εγκρίνεται. πίπτη 255, 256 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να σηκώνετε το χέρι όμω, διαφορετικά είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 123 άρτη ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 257, 265D υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 266D υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 143 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 258, 259 τώρα υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 259 άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρασε. απορρίπτεται. 185 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 267 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 268 δι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 204 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 269 δι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 206 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 270 D με ονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 208 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 271 D υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 219 υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 219 άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 272 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 273 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 228 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 31 έρθει ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 250, 42, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 251 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 260 δι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μονομαστική Κλίση Άρτη Ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ολοκληρώνεται κατά αυτόν τον τρόπο η πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έκθεση Φαγιών. 210 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία τη καθήλυνα αρμόδια επιτροπή από κοινού υπέρ κατά αποχέ εγκρίνονται. Τροπολογία 8 υπέρ παρακαλώ κατά αποχέ εγκρίνονται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 άρτη ψηφοφορία Πέρασε. εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος, άρθρη ψηφοφορία. Πέρασε. Γκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 114 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα τη 114, έτσι δεν είναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ. Μάλλον άρτη ψηφοφορία. Άρτη ψηφοφορία για την 146. Πέρας.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 Εγκρίνεται. 186. Άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 201. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 205 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 213 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 214 D υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 215 D υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 211 D υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 206 καταπίπτει, 216D τώρα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 164 υπέρ, κατά, αποχές, Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 164 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 207, 208 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 217 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 218 δι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 209 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται καταπίπτει 192, 212 D υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. Ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου με ονομαστική κλίση άρθρη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Η πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ολοκληρώνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Περνάμε στην έκθεση Χολμάιερ, Ταμείο Στερική ασφάλεια. Τροπολογία τη καθήλυνα αρμόδια επιτροπή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 1, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 8, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 11 πρώτο τμήμα άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Άρτη ψηφοφορία μάλλον. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50, πρώτο τμήμα. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 61 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Θέλετε να επαληθεύσουμε το δεύτερο τμήμα της 61. Πολύ ωραία. Άρτη ψηφοφορία λοιπόν. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 68. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. 71. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. 79. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 127 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 128 άρθρη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται 129 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 157 δι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 158 δι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Εγκρίθηκε 159, αλλά στο επαληθεύσουμε. άρθε ψηφοφορία για την τροπολογία 159. Πέρασε. Όντως εγκρίνεται. Τροπολογία 25, μάλλον αυτή καταπίπτει, 156 D υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 31 τώρα υπέρ, κατά, άποχε, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 31, άρτη ψηφοφορία παρακαλώ, πέρας. Εγκρίνεται ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου Μονομαστική κλίση. Άρτη ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Η πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ολοκληρώνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Περνάμε στην έκθεση Αγιούζο. Τροπολογία 195 Μονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ολοκληρώνεται έτσι. Περνάμε στην έκθεση Φέλκεν. Τροπολογία 6 με ονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται και ολοκληρώνεται έτσι και η πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περνάμε στην έκθεση Χάρκιν και Λάμπερτ. Τροπολογίες 1 με 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου. Μονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ολοκληρώνεται έτσι η πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περνάμε στην έκθεση Monte. Τροπολογία 10. Μονομαστική κλίση. Άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και ολοκληρώνεται έτσι και η πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περνάμε στην έκθεση Τέλιτσκα. Τροπολογία 18. Μονομαστική κλίση. Άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και ολοκληρώνεται έτσι και η πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για την έκθεση αυτή. Περνάμε εδώ πέρα στην έκθεση που έχει να κάνει με το Ταμείο για την Αλία και τις θαλάσσιες μεταφορές. Ο κύριος Κάντεκ έχει το λόγο, παρακαλώ. Ε, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ψηφίσουμε δύο επίγοντα μέτρα για την αλία. Για να είμαστε έτοιμοι, αν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ τη Ένωση και του Ηνωμένου Βασιλείου πριν τι 29 Μαρτίου τρέχοντο. Η Βουλή των Κοινοτήτων, όπω ξέρετε, απέρριψε την πρόταση τη ε, Τερέσα Μέη χθε το βράδυ. Υπενθυμίζω ότι τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν μόνο εάν υπάρξει αποχώρηση χωρί συμφωνία. Εάν, όπω ε, όλοι ή τουλάχιστον οι περισσότεροι επιθυμούμε υπάρξει συμφωνία, η Συμφωνία ε, Ελευθέρου Εμπορίου ή Τελειοναϊκή τηλεοναϊκή ενωση θα πρέπει να βασιστεί σε μια αμοιβαία συμφωνία πρόσβαση στα ύδατα και στου πόρου όπω γίνεται σήμερα. Και αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Ε, εκφράζω την άποψη τη Επιτροπή Αλία που υπενθυμίζει αυτή τη θέση για τι μελλοντικέ σχέσει μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ηνωμένου Βασιλείου και σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε κύριε Κάντεκ. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 1 υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται. Το σύνολο τώρα του κειμένου μονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και ολοκληρώνεται έτσι και η πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διοδοτήσεις αλλιές, γελευτικά σκάφη, Επιτροπή Αλίας πάντα αρμόδια. Τροπολογία 1, μονομαστική κλίση, άρτη ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Η πρόταση της Επιτροπής τώρα. Μονομαστική κλίση, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου ολοκληρώνεται και για την έκθεση αυτή. Έκθεση τώρα Ερτούγκ. Τροπολογία υπαριθμών 1, CP1, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 1, CP2. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου με ονομαστική κλίση. Άρτη ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Και ολοκληρώνεται κατά αυτόν τον τρόπο και η πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μια Ευρώπη που προστατεύει καθαρό αέρας για όλους. Ανθρωπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Μανομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Άχτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπίπτει το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Παράγραφος 4 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5 τώρα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 31 άρτη ψηφοφορία Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 μονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές. Να σηκώνετε τα χέρια όμως παρακαλώ πολύ. Ας παληθεύσουμε αυτή τη στιγμή την τροπολογία 10, άρτη ψηφοφορία, πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 16, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Παράγραφος 17 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 18 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα άρτη ψοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα άρτη ψοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. κάρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 15. Άρτη, ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Παράγραφος 28. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 24 τώρα. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 12. Πολύ ωραία. Άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρτη ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρασε. Όντως απορρίπτεται. Παράγραφος 35. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 13, άρτη ψηφοφορία, πέρας. Εγκρίνεται. 37. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 40 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ Ναι, ναι. 18 υπέρ. Μάλλον. Άρτη ψηφοφορία για τροπολογία 18. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 50 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται διορθώνει ο Πρόεδρος. Α το ελέγξουμε και ηλεκτρονικά τότε. Τροπολογία 14. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας, πέρας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 34 τώρα υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για 34 άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42. Μονομαστική κλίση. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 τώρα. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Άρτη ψηφοφορία μάλλον.